Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the next committee meeting. Let us take a seat. Καθίστε παρακαλώ. Να αρχίσουμε. Αν μπορείτε παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες σας στη σχισμή για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Παρακαλώ. Πατήστε το κουμπάκι. Τέλεια, πολύ ωραία δουλεύουν όλα. Πιλάρ, μπράβο. Λαμπρά. Ωραία. Θα ψηφίσουμε με την Πιλάρ. Η συνάδελφός μας, η κυρία Καηλή, δεν είναι έτοιμη ακόμη. Θα περιμένουμε λίγο. Εντάξει. <gasps> Εντάξει. Πατήσατε κόκκινο όμως. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Όλα λειτουργούν. Πρώτα θα ψηφίσουμε την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή. Προκλήσει, ευκαιρίε και διδάγματα για το σχεδιασμό πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητή μα, ο Ταμά Ντόιτ. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε και αυτήν ηλεκτρονικός. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Να την ελέγξουμε μια ακόμη φορά. <clears throat> Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε ηλεκτρονικός τροπολογία 58 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σύνολο των εγκεκριμένων τροπολογιών, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη. Πέρα της Καταπληκτικό αποτέλεσμα, 48 ψήφοι υπέρ, μία ψηφός κατά και τρεις αποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Όσον αφορά τώρα την ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 έως 2027, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη Συμφωνία. Ε, ήμουν εγώ εισηγητή του σχεδίου αυτού γνωμοδότηση. συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται, 3, υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται, 4, υπέρ, κατά, Έλεγχο. Δεν ήταν σαφέ για μένα το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικό στη 4. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Να την ελέγξουμε και αυτήν ηλεκτρονικός. Τροπολογία 5. Πέρασε. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 και 9 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, ψηφίζουμε την 58. Από τη 18 πηγαίνουμε στην 58. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος της τροπολογίας 58. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Προσθήκη συμβιβαστική 2. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, δύο προσθήκη που αυτή τη φορά ζητούν οι πράσινοι. Η προηγούμενη ήταν ε, αίτημα των σοσιαλδημοκρατών. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος μία ακόμη φορά. έλεγχος ε, της προσθήκης στη συμβιβαστική 2 που ζήτησαν οι πράσινοι. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Πάμε στη 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος της 17. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβιβαστική 3 που ζήτησαν οι πράσινοι. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος της προσθήκης στη συμβιβαστική 3. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος. Ελέγχουμε ηλεκτρονικό στην 24. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβιβαστική 4 που ζήτησαν οι πράσινοι. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρα στι ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβιβαστική 6 που ζήτησαν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες και οι πράσινοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Προσθήκη στη συμβιβαστική 8 που ζήτησαν οι πράσινοι υπέρ κατά Έλεγχο. Προσθήκη συμβιβαστική 8 που ζήτησαν οι πράσινοι. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά έλεγχος της 39 έλεγχος της τροπολογίας 39 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 35 υπέρ κατά Έλεγχος της 35. Έλεγχος της 35. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, έλεγχος. Έλεγχος της 63. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Της 65. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία στο σύνολο των τροπολογιών ε, που εγκρίθηκαν με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. And I close the Πέρας. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητηρία στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, δεν χρειάζεται να φύγετε. Γιατί έχουμε και το υπόλοιπο της ε, συνεδρίασής μας ε, για τις επόμενες δύο μισή ώρες. Είναι Πολύ σημαντικό αυτό να σας το πω, παρόλο που φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Let Ας πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, είναι το υπαριθμόν 11. Καθορισμός συγκεκριμένου χρηματοδοτικού 10 συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος για τον παροπλισμό ε, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Πίτερ Κουρουμπάσεφ και αφορά την αρρωγή προς τις χώρες οι οποίες πρέπει να ε, κλείσουν ε, πλέον το, τα ε, πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία πυρηνικά κέντρα, τα οποία έχουν φτάσει πλέον στο τέλος του κύκλου ζωής. Αυτό γίνεται βάσει του άρθρου 203. Αγαπητέ συνάδελφε Κουρουμπάζευ, αγαπητέ Πίτερ, έχετε το λόγο. Благодаря ви, господин председател. Агапите Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε ήδη, αυτά τα προγράμματα ε, παροπλισμού αφορούν, έχουν ήδη ενταθεί ε, στα προγράμματα ένταξης της Σλοβακίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν τον παραπλησμό των εγκαταστάσεων στο Κοσλοντούι και στο Μποχούνιτσε. Επομένως, η πρόταση αυτή ε, ε, αφορά τον παροπλισμό καθώς επίσης και τη διαχείριση των ε, αποβλήτων ε, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα επίσης του κοινού κέντρου έρευνας που αφορά και κέντρα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες. Μας ενδιαφέρει εδώ η διαχείριση όλων των ε, αποβλήτων, κυρίως δε των ραδιενεργών και το σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ε, μία κοινή δεξαμενή γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειριών ε, ο ρόλος του κοινού κέντρου έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό ε, ερευνητικό κέντρο, μια κοινή ερευνητική ομάδα η οποία θα συλλέγει ε, όλες τις ε, πληροφορίες και θα αποθυσαυρίζει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο διότι ξέρουμε ότι έχουμε πλέον διαδικασίες παροπλισμού σε διαφόρων, διαφόρων ειδών αντιδραστήρες σε πολλές χώρες εδώ μιλάμε όμως για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε φυσικά για αντιδραστήρες που βρίσκονται εντός της επικρατείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε τρίτες χώρες. Πρέπει ε, λοιπόν να ε, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προσαρμόσουμε τον 1368 Ευρατόμ ε, που, ε, και πώς να το εφαρμόσουμε στο Κοσλοντούι και στο Μποχούνιτσε. Ε, και να προσπαθήσουμε να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα με τη διαδικασία παροπλισμού της Ιγναλίνα. Ε, θα πρέπει να ε, δώσουμε την ε, δυνατότητα να έχουμε μία αντίδραση κοινή και ευρωπαϊκή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις και να αντιμετωπίσουμε σωστά τις προκλήσεις που δημιουργεί ή που έχει απέναντί της Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πυρηνικής ενέργειας. Οι προτάσεις αφορούν λοιπόν και την Σλοβακία και την Βουλγαρία ε, και ε, γίνεται μία πρόταση όσον αφορά ε, συγκεκριμένα ποσοστά. Βεβαίως εγώ μπορώ να μιλήσω κυρίως ε, για την χώρα μου, τη Βουλγαρία που την ξέρω καλύτερα. Χθες μιλήσαμε και για την περίπτωση της Ιγναλίνα ε, στην ε, Λιθουανία. Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε και ζητούμε μεγαλύτερη οικοδομική παρέμβαση από πλευρά της Κομισιόν τα όσα ε, προτείνονται αφορούν ε, και τα ποσοστά της χρηματοδότησης ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λόγος για ένα 50%. Εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο 50% ε, τώρα γίνεται λόγος για μια χρηματοδότηση της τάξης του 60% για τη Βουλγαρία και 63% για την ε, Σλοβακία. Ε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή η μείωση ε, της χρηματοδότησης για, τα, για τις δύο αυτές χώρες είναι σημαντική Πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη και τα χρονικά ε, περιθώρια. Για τη Βουλγαρία, ας πούμε, το χρονικό όριο είναι το έτος 2050. Αυτέ, με αυτά τα ποσοστά τα οποία προτείνονται δεν μπορεί να βοηθηθεί η χώρα έτσι ώστε ε, να ε, καταφέρει να φέρει σε πέρας την προσπάθεια. Μιλάμε εδώ για πλήρη παροπλισμό τεσσάρων αυτόνομων ε, ε, μονάδων, μπλοκ, για την Βουλγαρία έγινε λόγος ε, για πλήρη απενεργοποίηση των αντιδραστήρων που όμως είναι ακόμα λειτουργική. Και ε, καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες κοστίζουν και μάλιστα κοστίζουν πάρα πολύ. Κοστίζουν πάρα πολύ και όσον αφορά ε, την ε, ενέργεια και το, το κόστος της, της ενέργειας. Επίσης, να πούμε ότι στη Σλοβακία η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική γιατί οι αντιδραστήρες στη Σλοβακία είναι διαφορετικοί από τους αντιδραστήρες της, του Κοσλοντούι. Οπωσδήποτε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι διαδικασίες να είναι ε, αντίστοιχες με τον τύπο του αντιδραστήρα και επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εθνικές νομοθεσίες αλλά και ε, οι διαδικασίες και οι προσπάθειες που σε εθνικό επίπεδο έχουν ε, λάβει χώρα. Φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρήση η οποία γίνεται όσον αφορά τους αντιδραστήρες Εμεί αυτούς. Εμείς ζητούμε κυρίω στο σημείο 7 που αφορά την χρηματοδότηση, ζητούμε τροποποίηση. Να υπενθυμίσω ότι ε, οι εξελίξεις ε, στην Σλοβακία και στη Βουλγαρία μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ θετικό ε, προηγούμενο και οπωσδήποτε ε, εάν θέλουμε να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε ε, τον ε, παροπλισμό και την σταδιακή αποξύλωση όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων των διαφόρων χωρών. Αλλά οπωσδήποτε για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Οι σκιώδεις εισηγητές τώρα Εξ ονόματος του Έλκο Νέσβος Λάγγεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χτες μιλήσαμε για την Ιγναλίνα, η οποία έχει άλλη διάσταση από τις δύο αντιδραστήρες Βουλγαρίας-Σλοβακίας. Ε, η Ιγναλίνα στις διαπραγματεύσεις ένταξης έκλεισε. Θυμάμαι το 2006 και 2009 όπου οι αντιδραστήρε τύπου Τσερνομπίλ έκλεισαν. Στην περίπτωση Βουλγαρίας και Σλοβακίας, οι δύο αντιδραστήρες που συζητάμε, ε, συνεπάγονται πολύ μικρότερα προβλήματα. Πρώτον, τα προγράμματα διάλυσης έγιναν πολύ αποτελεσματικότερα, ταχύτερα, επιτυχέστερα, η τάξη μεγέθους είναι μικρότερη. Και δεύτερον, ε, σε αυτό το τομέα δεν χρειάζεται ε, να λάβουμε υπόψη μας ε, όσα διαπίστωσε ήδη το δικαστήριο το 2016 που συνέστησε υψηλότερη εθνική συνεισφορά κατά την περίοδο 2014-2020 και μετά το 2020 τα ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης θα σταματούσαν τα κράτη-μέλη θα έπαιζαν το ρόλο τους ε, αντιμετωπίζοντας ε, τα προβλήματα ε, με βάση την αρχή ορυπαίνων πληρώνει αλλά και τη διάθεση κονδυλίων για τον παραπλησμό. Τώρα πρόκειται για Κοσλουντού και Μποχουνίτσε, Σλοβακία-Βουλγαρία και ο συνάδελφος ασχολήθηκε με όλη αυτή τη θεματική. Γενικά συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Εκεί που έχω επιφυλάξεις, γιατί πρόκειται για το αντίθετο με την απόφαση του δικαστηρίου πριν από δύο χρόνια, είναι η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 50% στα 60%. Αυτό αντιβαίνει στις μέχρι τούδε προσπάθειές μας. Το ίδιο αφορά και την Ιγναλίνα. Εκεί είχαμε 20% και η εισηγήτρια πρότεινε μόνο 14%. Τα 86% συγχρηματοδότηση ε, πρέπει να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φαίνεται με πρώτη ματιά απλό, αλλά γενικά με βάση την πολιετή μου πείρα η πιο αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων ε, παροκλισμού ε, πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή του κράτους μέλους και διότι θα πρέπει να έχει ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο κράτος μέλος για τον παροπλισμό. Αυτό πρέπει να το δούμε. επίση, να δούμε και κάτι άλλο. Το κοινό κέντρο έρευνας στο Βέλγιο, Ίσπρα και Ολλανδία, Ιταλία και Ολλανδία και στην Καλσρούη. Αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους. Ε, αποθήκευση δηλαδή ε, έχει νόημα να γίνεται εκεί, συμφωνώ εδώ με τον εισηγητή, αλλά από την άλλη πλευρά αν σκεφτώ τη γενικότερη κατάσταση της πυρηνικής ενέργειας, το, τα μισά κράτη-μέλη κάνουν ή κάνουν νέε ε, ε, ε, κατασκευές ε, ή μικρές μονάδες. Ενώ στη χώρα μου, τη Γερμανία, τα πυρηνικά εργοστάσια θα πρέπει να κλείσουν μέχρι το 2022 χωρίς ενωσιακά κονδύλια. Και στη δική μου εκλογική περιφέρεια το νεότερο εργοστάσιο ε, που κατασκευάστηκε το 88 κλείνει τώρα χωρίς καμία ευρωπαϊκή συμμετοχή. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει το ποσοστό που συμφωνήθηκε να διατηρηθεί, αλλά να δούμε ε, και να φροντίσουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύντομα. Ε, νομίζω ότι σε αυτά θα διατηρήσουμε τη διαφορετική μας γνώμη. Για την ομάδα EFDD, όχι ο κύριος ε, Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους Σκιώδης για την ε, διεξοδική εξέταση των προβλημάτων και την παρουσίασή τους εδώ. Μιλάμε για προβλήματα σε πυρηνικά εργοστάσια που καμιά φορά βρέθηκαν αντιμέτωπα με παράδοξες πολιτικές αποφάσεις. Ε, ε, κάποια συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το 2017 χωρίς πρόβλημα. Ο εισηγητής το ανέφερε ήδη αυτό. Πρέπει επίσης να σας πω ότι σήμερα προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες ότι προσπαθούμε να κλείσουμε πυρηνικά ε, εργοστάσια, όχι συνήθεια εργοστάσια και συνήθεις εταιρείε. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τους δικούς μας χρηματοδοτικούς πόρους. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι ένα ελάχιστο ποσό πρέπει να τεθεί για την ενωσιακή χρηματοδότηση και μετά θα πρέπει το ποσό αυτό να αυξάνεται ε, σε συνδυασμό με την ταχύτητα των δράσεων παροπλισμού, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο. Επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιτροπή, ένα κέντρο έρευνας, το οποίο θα συλλέγει εμπειρία παροπλισμού από τις διάφορες χώρες και μετά θα ε, γίνεται επιμερισμός της εμπειρίας σε νοσιακά και μη νοσιακά όργανα. Αυτό θα δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάσιμο Γκαρίπα από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχήν ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κουρουμπάσεφ, για το εξαιρετικό έργο του κατά την εξέταση της πρότασης. Συζητήσαμε και χθες στην ίδια Επιτροπή την περίπτωση Ιγναλίνα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτήν. Θα επικεντρωθώ στην ε, συγκεκριμένη πρόταση. Να θυμίσω δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι κέρια προτεραιότητα της Ένωσης και γι' αυτό η Κομισιόν υπέβαλε την πρόταση αυτή για να οριστικοποιήσει τον παροπλισμό των δυο, Κοσλοντούι και ε, Μποχουνίτσα. Το δεύτερο στρατηγική σημασίας ε, ζήτημα που ανακύπτει εν προκειμένου είναι ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ο παροπλισμός Κοσλοντούι, Μποχούνιτσε και του Κοινού Κέντρου Έρευνας ε, που είναι της Κομισιόν. Γιατί, Γιατί θεωρήθηκε αναγκαίο η, η, διαμήραση πληροφοριών και γνώσεων θα προωθήσουν αυτή την προηγμένη φάση του παροπλισμού. Συμφωνώ απόλυτα εν προκειμένου με τις παρατηρήσεις του εισηγητή. Να πω ακόμα ότι τα ποσά που αναφέρονται στις προτάσεις της Κομισιόν είναι εκείνα που είναι στο σχεδιασμό παροπλισμού για τις δύο χώρες, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία. Και θεωρούνται απόλυτα αναγκαί, ε, ικανά για να ολοκληρωθούν οι ε, παροπλισμοί το 2025 και το 2030 αντίστοιχα. Και προχωρούμε τώρα στο τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω για τις πρακτικές συγχρηματοδότησης. Η συγχρηματοδότηση στις δύο χώρες είναι μεταξύ 30 και 40%. Και, όπως είπε και ένα αξιότιμο μέλος, κατά την παρέμβασή του, το 2016 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι η αυξημένη συμμετοχή από τον δικαιούχο αυξάνε, αυξάνει την διαδικασία οικειοποίησης του ιδίου του έργου. Γι' αυτό η Κομισιόν θεώρησε σωστό να αυξήσει το ποσοστό τη προτινόμενης χρηματοδότηση από, από το κράτος μέλος και να περιορίσει τη δική της συμμετοχή στο μέγιστο του 50%. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοχίτσεφ, κυρία Δεσεβαλιέ, δεν μας ε, είπατε ότι ζητείτε το λόγο και δεν η, η κυρία Σεβαλιέ είναι σκιώδης. Αλλά η Ρώμη δεν είναι στο κατάλογο. Πάντως έχει το λόγο ως εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, απλός μηχανικός είμαι δεν είμαι ειδικό ε, στην ε, πολιτική, γι' αυτό ε, ακριβώς δεν ζήτησα να ε, είμαι εισηγητής, ε, δεν είμαι εισηγητής. Ε, θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ γνωρίζω από τη χώρα μου την κατάσταση και θα ήθελα να πω προς τον εισηγητή ότι πρέπει να γίνει παροπλισμός βάσει κυβερνητικής απόφασης όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων που πρέπει να παροπλιστούν. Είναι δική τους απόφαση, η χρηματοδότηση είναι δική τους. Όμως η Συμφωνία Προσχώρησης Τριών Κρατών τριών κρατών της Λιθουανίας, της Βουλγαρίας και της Σλοβακίας συμπεριλαμβάνουν τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων που είναι επιβεβλημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συνεισφέρουμε στον παροπλισμό αυτό και μου κάνει εντύπωση που κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει καμία τεχνική γνώση αποφασίζει την αύξηση της συμμετοχής της κάθε ε, μιας από τις χώρες αυτές. Θα ήθελα να καλέσω τους εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια τεχνική συζήτηση ξέρουν ποιο είναι, ποιος είναι ο όγκος τσιμέντου που πρέπει να απομακρύνουμε, τι ακτινοβολία υπάρχει ε, στην εγκατάσταση σε κάθε είδος υλικού, πώς να διαχειριστούμε το χάλιβα και το... Το τα σύνθετα υλικά ειδικότερα στη Λιθουανία υπάρχει και μία ακτίνα 10 χιλιόμετρων ε, γύρω από την ίδια την εγκατάσταση Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ποτέ παροπλήσει εσείς στο παρελθόν κάποιο τέτοιο, είδο, κάποιο τέτοιο είδους ε, εγκατάσταση. Κάτι ξέρω εγώ σχετικά με αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα, ε, τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Χτες μιλούσαμε γενικότερα για τα προγράμματα, για το μέλλον, για την επιθεώρηση, την διαχείριση διαφόρων ε, ραδιενεργών υλικών, είτε χαμηλής είτε υψηλής ακτινοβολίας ε, και την χρήση αυτών των υλικών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συμπεριλάβουμε στα προγράμματά μας ε, γιατί τώρα συζητούμε για δεκάδες αντιδραστήρες στη Γερμανία, για τους αντιδραστήρες αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκθεση. Όμως υπάρχουν και άλλοι μικροί αντιδραστήρες, για παράδειγμα στο κέντρο της ε, Βιέννης, στο πανεπιστήμιο τους. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα χρειαστεί να παροπληστεί και αυτός, όπως και οι αντιδραστήρε που συζητούμε σήμερα. Είμαι σίγουρο ότι σε, πολλούς, σε πολλά πανεπιστήμια υπάρχουν μικροί αντιδραστήρε και αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τι θα κάνουμε με το υλικό των συγκεκριμένων αντιδραστήρων πώς θα διαχειριστούμε τα ραδιενεργά υλικά χαμηλής και υψηλής ραδιενέργειας, ακτινοβολίας και είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει και στην Αυστρία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα ούτω ώστε να διευκολυνθεί η επίλυση αυτού του προβλήματος και φαντάζομαι ότι ο κύριος Λάγκεν θα συμφωνήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λουσεφαλία. εκ μέρους της ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι σημαντικό να, υπάρχει χρήμα, να υπάρξει χρηματοδότηση του παροπλισμού και της διάλυσης των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και των αντιδραστήρων. Μόνο τρεις έχουν ε, αυτή τη στιγμή παροπληστεί. μόνο πέντε ε, λειτουργούν σε, ολόκληρο τη Γαλλία, σε ολόκληρη τη Γαλλία, κάτι που είναι μια τεράστια πρόκληση. Η διάλυση των, πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Βουλγαρία και στη Λιθουανία είναι κάτι το οποίο ήταν ε, γραμμένο στην ε, συνθήκη προσχώρησής τους, επομένω είναι κάτι που πρέπει να τύχει σεβασμό. Τα 14 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα οποία αφορά, πρέπει να μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις τους, αλλά και, και για την χρήση των υλικών, αλλά και για την διαχείριση των αποβλήτων. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη διαχείριση για το μέλλον, για όλα τα κράτη-μέλη στο μέλλον. Το JRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις πολιτικές κατευθύνσεις που θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση η το ενεργειακό μείγμα δεν πρέπει να προέρχεται από ε, ιδεολογίες αλλά από την ελεύθερη βούληση των κρατών μελών. Η Βουλγαρία και η Λιθουανία έχουν χάσει μεγάλα εισοδήματα λόγω της, ε, του κλεισίματος των αντιδραστήρων αυτών. Εδώ και πολλά χρόνια πρέπει να τις συνοδεύσουμε, να τις βοηθήσουμε, ειδικά όταν υπάρχουν ε, ζητήματα ασφαλείας. Όλοι θα κερδίσουμε σε εμπειρία, όμως δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει στις στρατηγικές επιλογές των κρατών μελών. Φαίνεται λογικό να υπάρχει ένα και μόνο πρόγραμμα κοινό ώστε να ε, υπάρχει μια συγκέντρωση πόρων και διευκόλυνση ε, της ε, διάλυσης των εγκαταστάσεων. Νομίζω όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, για να μην υπάρχει αποποίηση ευθυνών από πλευράς των κρατών μέλων. Νομίζω ότι η συγχρηματοδότηση 50% είναι μια καλή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάγκεν, θα σας δώσω το λόγο γιατί δύο φορές ε, σας ανέφερε ο συνάδελφος. Σας δίνω το, το λόγο για ένα λεπτό. Είναι ζωντανή η συζήτηση, γι' αυτό ξαναζητώ το λόγο. Ο συνάδελφος μηχανικός και αντιπρόεδρος είπε ότι από το θέμα από δεν, ε, δεν το ξέρει σε πολιτικό αλλά σε τεχνικό επίπεδο. Μέσα από το πρίσμα της ε, τεχνολογίας ε, δεν θέλει να περιορίσει κάτι. Εμείς είπαμε ότι για τη Λιθουανία το συνολικό κόστος θα είναι 1,5 δις ευρώ, εκεί εκτιμώνται, για τη Βουλγαρία 731 εκατομμύρια, για τη Σλοβακία 671 εκατομμύρια, 890 εκατομμύρια για την έρευνα των επιπτώσεων, Οπότε ε, είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Συνολικά ε, έχουμε 8 αντιδραστήρες ε, παλιάς γενιάς σοβιετικής κατασκευής. Αυτό ήταν το κλείσιμο προϋπόθεση για να μπουν οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ήταν και κατάλληλη χρηματοδότηση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η το 2008, θυμάμαι, ήταν ακριβώς πριν από 10 χρόνια όταν ο Ρώσος ε, μηχανικός και επικεφαλής της επιχείρησης του εργοστασίου είπε ότι έχετε επενδύσει 300 εκατομμύρια για την αναβάθμιση της ασφάλειας. Παλιότερα είχαμε 30 με 40 ε, σοβαρά ατυχήματα ανά έτος. Σήμερα δεν έχουμε κανένα ατύχημα και παρόλα αυτά πρέπει να, να κλείσει το εργοστάσιο. Τώρα οι προϋποθέσεις είναι, ε, αυτε, εδώ οι προϋποθέσεις είναι τελείως διαφορετικές. Γι' αυτό στην περίπτωση της Ιγναλίνα μπορούμε με ε, ήσυχη συνείδηση να δώσουμε 80% στους άλλους 50%. Είναι σωστός ο συντελεστής το ποσοστό. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί περαιτέρω αύξηση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν ερωτάτε αν ε, έχει κάποιο πολύ σύντομο σχόλιο. Σύντομα γιατί μετά τις ομιλίες θα είναι το δεύτερο, η δεύτερη παρέμβασή σας. Ο κύριος Μάσιμο Γκαρίμπα. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχω λόγο να σχολιάσω. Πάρα πολύ ωραία. Πίτερ Κολομπάσεφ. Έχετε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια των σκιωδών. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Βουλγαρία ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ζητήσει από την ε, Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Λιθουανία να παροπλήσει τις ε, πυρηνικές εγκαταστάσεις εν είδη, ε, εν είδη τηλεσυγράφου. Και ε, ξέρετε, δεν ήταν απόφαση που ελήφθη από κυρίαρχη απόφαση από μια κυρίαρχη χώρα ε, ε, ε, πρόκειτο για μία απόφαση την οποία επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξεκίνησε τις συζητήσεις με τις νέες χώρες. Μία από τις προϋποθέσεις των ουκάνεφε ήταν ακριβώς αυτός ο παραπλησμός των αντιδραστήρων. Όπως είπε άλλωστε και ένας συνάδελφος πριν, ο αντιδραστήρας ε, της ε, ε, Λιθουανίας, όπως άλλωστε και η δική μας στη Βουλγαρία, είναι ακόμα λειτουργική. Εμείς έχουμε λάβει βοήθεια πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ για μία περίοδο 7 ετών και είναι γεγονός ότι εμείς προσπαθήσαμε τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πάντως στην Κομισιόν ότι οι δεσμεύσει, το επαναλαμβάνω, επευλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τελεσίγραφο. Δεν είχαμε δυνατότητα να ε, ε, μην το δεχτούμε αν θέλαμε να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επρόκειτο, επαναλαμβάνω, για κυρίαρχη απόφαση από κυρίαρχους λαούς. Βεβαίως, εμείς έχουμε πλέον ε, την ευθύνη αυτών των αντιδραστήρων και εμείς έχουμε την ευθύνη για το τι θα συμβεί αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε για μείωση της ε, χρηματοδοτικής παρέμβασης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία και η Σλοβακία, χώρες για τις οποίες γίνεται λόγος εδώ στη συγκεκριμένη ε, έκθεση, μπορούν να αποτελέσουν ε, παράδειγμα γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ πρόβλημα σε αυτούς τους αντιδραστήρες που λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο. Επομένως, ε, ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε μόνο θετικές εμπειρίες. Να μην λησμονούμε ότι υπάρχει και το κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και εκεί ζητώ να δημιουργηθεί και μια κοινή ομάδα ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών, εκπόνησης καταλήλων μέτρων κλπ. Όλα αυτά να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες 18 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Ήτρε και ψηφοφορία ε, στην Ήτρε 3 Δεκεμβρίου. Έχουμε τώρα το επόμενο θέμα, κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση για το ΙΤΕΡ και ανάπτυξη πυρηνικής σύνδεξης. Εξαιρετικό, ε, εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Πρόκειται για μια διεθνή ε, κοινοπραξία έχουμε τον συνάδελφο Μαρινέσκου, ο οποίος είναι εισηγητής. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι σε αυτή την περίπτωση ε, δεν είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν να διαβουλευτεί το Κοινοβούλιο. Ε, ωστόσο, το Κοινοβούλιο αποφάσισε λόγω της σημασίας ε, του θέματος να εκφραστεί μέσω εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας. Έχουμε συζητήσει το θέμα επανειλημμένα και εδώ έχουμε την απάντησή μας προς την πρόταση της Κομισιόν ε, που αφορά την τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου μέσω της οποίας ε, τροποποιείται ε, η απόφαση 2007-198 Εδώ μιλάμε ε, για πολλά χρήματα και επομένως είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όσοι εισηγητής ο κύριος Μαριάννο Μαρινέσκου θα έχει το λόγο για μερικά, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ίτερ είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε. Ε, το τελευταίο καιρό το project προχωράει ε, με ταχύ ρυθμό. Δεν υπάρχουν πλέον τα προβλήματα τα οποία ε, υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχει τώρα και έχει γίνει, μάλλον έχει ολοκληρωθεί μια εξωτερική, ένας εξωτερικός οικονομικός έλεγχος που δείχνει ότι μπορεί να προχωρήσει το έργο. Εγώ ασχολούμαι με διοικητικά ζητήματα κιόλα στην γνωμοδότησή μου. Διότι υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα όσον αφορά συγκεκριμένες ε, ε, διοικητικές και χειριστικές επιτροπές. Δεν γνωρίζουμε ας πούμε τον ακριβή αριθμό των μελών τους ή κάθε πότε πρέπει να συνεδριάζουν. Κατά τα λοιπά μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητέ συνάδελφε, είσαστε σύντομος και σαφής. Ε, και πολύ αποφασιστικός στα όσα μας είπατε και στην πρότασή σας. Ο κύριος Τζανονάτο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, με το οποίο μπορώ σε μεγάλο βαθμό να συμφωνήσω. Ε, κυρίως συμφωνώ με την ε, αναφορά του για την κατάλληλη χρηματοδότηση του τομέα της έρευνας καθώς επίσης και την ευχή να αποδείξει το ίτερ, ο οργανισμός ίτερ στο μέλλον ότι η σύνδεξη μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα αποτελέσματα. Ε, μπορούμε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε την σύνδεξη ε, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μίας ώρας τουλάχιστον. Οπωσδήποτε συμμερίζομαι και με τον εισηγητή ε, τα όσα αναφέρει όσον αφορά το προπολογισμό έτσι ώστε το επόμενο ΠΔΠ να λάβει υπόψη τι, το ύψος της απαραίτητης χρηματοδότησης της Ευρώπης μαζί με τις άλλες χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν. Επίσης, θεωρώ ε, σκόπιμη ιδιαίτερο ε, στην παράγραφο ε, στην οποία καλεί το Συμβούλιο να περιλάβει διατάξεις οι οποίες να δημιουργούν συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ ΙΤΕΡ και Προγράμματος Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ευρατμόμ για την περίοδο 2021-2023. Επίσης, το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική αυτή την αναφορά στην εκτίμηση της συμβολής ε, σε ε, είδος. Ε, και επίσης συμφωνώ με τα όσα αναφέρει σχετικά με τη Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή, Επιτροπή Προμηθειών και Συμβάσεων, τη σύνθεσή τους, προσωρινό ή μόνιμο καθεστώς κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ε, επίσης ε, συμφωνώ με ε, αυτό που λέει ο εισηγητής σχετικά με το κράτος υποδοχής αλλά νομίζω ότι εδώ χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες όσον αφορά το θέμα αυτό και το σημείο αυτό. Επίσης, όπως και στην ανακοίνωση 319 του 2017 της Κομισιόν, ε, ε, νομίζουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, κοινή αντιμετώπιση του θέματος έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και το χρονοδιάγραμμα θα γίνει δεκτό. Θα ε, ενθαρρύνουμε επίσης ε, την ε, Κομισιόν να ζητήσει περαιτέρω διαλεύκανση ορισμένων σημείων. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαβούλευσης του Κοινοβουλίου από πλευρά του Συμβουλίου. Επίσης θα υπάρχει επομένως μια δικιά μου τροπολογία που ε, θα ε, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει ενδεχόμενη τροποποίηση της συνθήκης Ευρατόμου που θα προβλέπει και την ε, διαβούλευση με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να δώσει το Κοινοβούλιο τον σαφή νομοθετικό του ρόλο. Τέλος, να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς επιστημονικής και ερευνητικής, όπου συμμετέχουν 7 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν με τρόπο πολύ ικανοποιητικό για ένα θέμα το οποίο και ένα ε, ε, ε, θέμα λοιπόν και ένα πρόγραμμα το οποίο από άποψη εμπειρική είναι πάρα πολύ σημαντική. σημαντικό. θα πρέπει να αποφύγουμε ε, ε, ε, τροποποίηση των προτινομένων και τροποποίηση επίσης του χρηματοδοτικού κόστους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό το σχέδιο ιτέρ, όταν βλέπω την τροπολογία του αγαπητού συναδέλφου εισηγητή, λέει ότι ο ΙΤΕΡ θα λύσει το πρόβλημα της ε, θέρμανσης ε, του πλανήτη. Θα ήθελα να σας πω ότι η θέρμανση του πλανήτη, αν είμαστε στο 2050 και έχουμε φτάσει στο συν, σε 3 βαθμούς, είναι πολύ αργά. Αν είμαστε στο 2100 και έχουμε επιπλέον 4 ή 5 βαθμούς, πάλι πολύ αργά θα είναι. Όταν λέμε λοιπόν ότι η σύνδεξη θα έπρεπε να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί είναι κάτι το οποίο ε, είναι ανεξάντλητο και ότι συνάδει με την περιβαλλοντική και ανταγωνιστική μας πολιτική κλπ. κλπ. Νομίζω ότι το παρακάνετε, γιατί όταν λέμε ανταγωνιστικό, δείτε για παράδειγμα ε, τι έγινε με τον ΙΤΕΡ. Ήμασταν στα 5,9 δις, τώρα είμαστε στα 19 δις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας είπε 65 εκατομμύρια δολάρια ε, θα θα διαθέσει ε, για το ίδιο θέμα. Εμείς όλο προσθέτουμε σε αυτόν τον προπολογισμό. Συνεχώς λέμε ότι πρέπει να περικόπτουμε το, το κόστος, αλλά στο ΙΤΕΡ είναι η Ευρώπη, είναι τα διάφορα κράτη-μέλη, ο καθένα συνεισφέρει για ένα συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού και βλέπουμε ότι οι ανισότητες είναι πάρα πολύ μεγάλε. υπάρχει και ένα ζήτημα τεχνικό. Ε, μιλάμε για ε, ε, εκατοντάδες, για εκατομμύρια ε, βαθμούς Κελσίου και δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της, του, της οικοδόμησης αυτού του, του κτηρίου. Εσείς πότε πιστεύετε ότι ο, ο ΙΤΕΡ θα συνδεθεί με την ηλεκτροδότηση ε, γιατί μόνο το πλάσμα θα ε, κατασκευάζει, μετά θα υπάρχει ένας δεύτερος αντιδραστήρας και μετά ένας τρίτος που θα είναι ο αντιδραστήρας παραγωγής, αλλά ο ΙΤΕΡ δεν θα παράγει ε, ηλεκτροδότηση. Είχαμε πει 2050, αλλά επειδή 10 χρόνια έχουμε ήδη καθυστερήσει, τελικά τι επίπεδο στόχου θα επιτύχουμε. Το θέμα λοιπόν ε, του κόστους ε, διάλυσης του ΙΤΕΡ το έχουμε συμπεριλάβει. Το 2010 το είχαμε πει θα το συζητήσουμε. Πού έχουμε φτάσει ως τώρα είναι, έχουμε τη σύνδεξη. Γνωρίζω πολύ καλά τη ραδιενέργεια, ε, γιατί έχω ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Ε, ε, είναι ένα ραδιενεργό υδρογόνο. Αν ποτέ γίνει ατύχημα, θα υπάρξει, θα εκλειθεί παντού ε, αυτή η ε, ουσία. Σε επίπεδο μετάλλων, για παράδειγμα, κάθε φορά που κάνουμε ακτινοβόληση ε, για να επιτύχουμε σύνδεξη υπάρχει όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερα αργενικά απόβλητα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι κατά τη γνώμη μου το ΙΤΕΡ είναι η μεγαλύτερη κατασπατάληση ευρωπαϊκού Χρήματο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Όλοι λέμε είναι κατεπήγον, περιβάλλον κλπ. Αλλά αυτό το θέμα του ΙΤΕΡ δεν θα μα βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημά μα. Αυτά ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι και θα ήθελα να συμφωνήσω με, αυτό που είπε ο συνάδελφο προηγουμένω. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την Ευρατόμ, γιατί εμεί μία, μία γνώμη απλώ εκφράζουμε δεν ε, μας δίνουν και πολύ σημασία. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει επιτέλους μια αναθεώρηση της συνθήκης αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Κοχίτσεκ, ο μηχανικός μας, ε, θα λάβει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας. Έχουμε συζητήσει πολύ και χθε μάλιστα για το μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα και πρόγραμμα ανάπτυξης και είπαμε ότι τα προγράμματα πρέπει να είναι προγράμματα εχμής. Και το πρόγραμμα σύνδεξης είναι ένα ε, πρόγραμμα Εχμή, Μιλήσατε για τις υψηλές θερμοκρασίες, μιλήσατε για ένα περιβάλλον εντελώς άγνωστο σήμερα. Κατασκευάζουμε το πλάσμα μέσα σε αυτούς τους αντιδραστήρες. Στον ιτέρ του σήμερα κατασκευάζουμε ε, το πλάσμα και πρέπει κάπως να το συμπυκνώσουμε. Αυτό είναι το πρώτο μας πρόβλημα. Βέβαια, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος της θέρμανσης του πλανήτη, για παράδειγμα. Σε ένα δεύτερο στάδιο, όπως είπατε κι εσείς, θα υπάρχει μια δοκιμαστική ε, εγκατάσταση και σε μια τρίτη φάση, ελπίζω να ζουν τα παιδιά μας ε, ακόμη, ε, θα είμαστε σε θέση να παράγουμε ενέργεια. Αυτό είναι το σχέδιο. Είναι έρευνα αιχμή αυτή. Και δεν μπορούμε να πούμε εκ των προτέρων αν η κατεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε είναι η σωστή. Έτσι γίνεται στην έρευνα. Παρ' όλα αυτά είναι έρευνα εχμής είναι κάτι το εντελώς μοναδικό και πρέπει προφανώς να αναρωτηθούμε για αυτά που είπατε. Τι να κάνουμε με τα υλικά όταν θα χρειαστεί να... Ε, ε, διαλύσουμε όλη αυτή την εγκατάσταση Πράγματι, όλα αυτά πρέπει να μα απασχολήσουν, Όμω πρόκειται για έρευνα αιχμή. Γι' αυτό πρέπει να την υποστηρίξουμε, κατά τη γνώμη μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένα ε, εμπορικό σύλλογο. Ε, δεν αφορά μόνο την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, αλλά και των ιδεών. Η έρευνα αιχμή, λοιπόν, είναι κάτι που μπορεί να μα επιτρέψει να διατηρήσουμε την ηγετική μα θέση στον κόσμο. Η ΤΕΡ είναι τμήμα αυτή τη προσπάθεια, γι' αυτό τον υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ταμπουράνο είναι ο επόμενος ομιλητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο για τα όσα ε, έχει αναφέρει σχετικά με την ε, προσπάθεια προώθησης ε, του ρόλου του Διεθνούς Οργανισμού Ίτερε. Αν συμφωνούσαμε με την αρχή θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και τον συνάδελφο. συμφωνούμε πάντως με τον συνάδελφο Τζανάτοβο ότι οπωσδήποτε θα πρέπει ο ρόλος του Κοινοβουλίου να είναι σημαντικός και να έχει λόγο όσον αφορά και το Ίτερε αλλά και άλλα θέματα. Ε, όσον αφορά το ίτερ, ε, ε, εμείς έχουμε θέση αμφιβολίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Όχι γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντική η διαρεύνηση άλλων πεδίων όσον αφορά την έρευνα και την πρόοδο, αλλά αυτά τα χρήματα, αυτά τα ατελείωτα ποσά δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εδώ. Χρησιμοποιώντας την πρώτη φράση ε, ότι η σύνταξη θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στο, στο καινούριο πεδίο της, στο, στο καινούριο πεδίο της έρευνας. Ε, κοιτάξτε, εδώ και ε, σχετικά με το Παγκόσμιο Μελλοντικό Ευρωπαϊκό και Ενεργειακό Τοπίο, Δυνητική Ανεξάρτητη, Ασφαλή, Φιλική προ το Περιβάλλον και Οικονομικά Ανταγωνιστική Πηγή Ενέργεια, αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημά μα, γιατί θεωρούμε ε, ότι ε, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τόσα πολλά χρήματα από του πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και των χωρών ε, για κάτι το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να είναι ασφαλέ και, και φιλικό, αλλά που για την ώρα δεν μα έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Ε, ε, ε, εάν πραγματικά είχαμε αφήσει την πυρηνική ενέργεια να αναπτυχθεί, ίσως να είχε καταστραφεί όλη η ανθρωπότητα. Επίσης, εδώ μιλάμε για, το, για έναν, για συγγνώμη, χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2030, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε την ανθρωπότητα από την κλιματική αλληλεγγύη κλπ. Σήμερα θα πρέπει πραγματικά να γίνει η διαφορά μέσα από χρηματοδότηση ε, των ε, πραγματικά καθαρών μορφών ενέργεια, των αναλλακτικών δηλαδή μορφών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ε, επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, ε, τα διασυνδεδεμένα δίκτυα, να προωθήσουμε άλλε μορφές ε, μετακίνηση. Δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν, δεν είναι δυνατόν να καθυστερούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε και τελειώνουμε με μια φιλοσοφική νότα γιατί ίσως θα πρέπει να περάσουμε και πέρα από τα τεχνοκρατικά. Η ανθρωπότητα είναι αρκετά σοφή έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τις ενέργειες, τους διάφορες μεφρές ενέργεια. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεσοβαλία ήταν η επόμενη, αλλά δεν βλέπω να είναι εδώ. Επομένω. η κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ε, συγχαρώ τον συνάδελφο Μαριάν Μαρινέσκο, τον συνάδελφό μας, για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Ε, θα υπενθυμίσω ότι ε, ο ΙΤΕΡ δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνές πρόγραμμα και αφορά την δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλες χώρες από ολόκληρο τον κόσμο. Και το πλεονέκτημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τον ΙΤΕΡ στην επικράτειά της, στο έδαφος της ρώτησε ε, και βεβαίως αυτή η χρηματοδότηση ε, του ύψους του 45% είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά δεν είναι δυνατόν ε, άμεσα να συλλέξουμε κατά κάποιο τρόπο, να δράξουμε τους καρπούς του προγράμματος αυτού, το οποίο αφορά κυρίως τις μελλοντικέ γενιές και εμείς σαν πολιτικοί θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια στιγμή τις μελλοντικέ γενιές. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι ένα περίπλοκο σχέδιο, ναι, είναι γεγονός ότι είναι ένα δύσκολο ε, στη διαχείρισή του ε, σχέδιο γιατί ακριβώς έχει αυτή την ε, διεθνή μορφή. Ωστόσο είναι πάρα πολύ θετικό όχι μονάχα για την ενέργεια σύνδεξης που είναι πολύ σημαντική από άποψη ερευνητική αλλά είναι και ένα project το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις τις οποίες δεν έχουμε σήμερα. Επομένως είναι σημαντικό να επενδύσουμε στον τομέα αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε απόλυτα να καινοτομήσουμε, κυρίως δε ή και πολλό δε μάλλον που αυτές οι καινοτομίες ε, μπορεί να έχουν επίπτωση σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Επομένως ε, δεν αφορά μονάχα τη σύνδεξη το θέμα αυτό, έστω και αν η σύνδεξη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα από μόνο του αλλά ε, ακριβώς μπορεί να δημιουργήσει νέες γνώσεις ε, αυτό το πρόγραμμα ITER ε, ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας. Ναι, φυσικά, φυσικά το ένα δεν αναιρεί το άλλο και κάνουμε ένα σωρό προσπάθειες και προς αυτήν την ε, ε, κατεύθυνση. Εδώ μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν. Μιλάμε για θέματα μη συγκρίσιμα. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ και συμφωνώ με το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Μούντ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδες. Μετά από τα σχόλια άλλων συναδέλφων, πρέπει να πω ότι το έργο είναι εντυπωσιακό και σημαντικό, κάτι που πρέπει να το αξιολογεί πάρα πολύ ε, θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί επηρεάζει τις αλλαγές στο κλίμα και αν δεν ανταποκριθούμε εκεί παραμελούμε τις υποχρεώσεις μας. Είναι ζωτικό αυτό το θαραλέο πρόγραμμα να είναι μέρος της απάντησής μας στην κλιματική αλλαγή και σε άλλες τεχνολογικές προκλήσεις. Επίση, ήδη αποδίδει για τους Ευρωπαίους πολίτες αποδίδει ε, σε τεχνολογία εχμής, αν δούμε δηλαδή την ε, τηλεδιαχείριση και τα νέα υλικά που προκύπτουν από αυτό το πρόγραμμα. Και όπως είπαν και άλλοι, είναι και διεθνές, με μια μοναδικότητα στην κλίμακά του. Και εμείς ε, είμαστε, έχουμε ηγετικό ρόλο και σε ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει αυτό το σημαντικό έργο. Και τελειώνω με αυτή τη διεθνή διάσταση, γιατί ένα μια σημαντική συνιστόσα στο πρόγραμμα αυτό ε, είναι η κοινή ευρωπαϊκή ε, διάσταση που μπορεί να προσφέρει στην ε, ε, ανάπτυξη το 2025. Και αυτό θέλω να περιγραφεί και να τονιστεί στο έργο αυτό. Thank you. Thank you Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Η κυρία Λεσεβαλιέ Ζητεί το λόγο, θέλετε. Όχι, ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ο κύριος Μάσιμο Γκαρίμπα. Ευχαριστώ, πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή νομίζω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Σχολιάζοντας την πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω, όπως είπε και εκείνος, ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχόλια ήταν διοικητικής φύσεως, αλλά σημαντικά κατά τη γνώμη μου για να στηρίξουμε και να διευκρινίσουμε την πρόταση. Η Κομισιόν λοιπόν θα δει τις προτάσεις αυτές πολύ προσεκτικά. Ακούγοντας τώρα τα σχόλια των διαφόρων μελών, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο ΙΤΕΡ είναι ένα πρόγραμμα διεθνές ε, μακροπρόθεσμο και πολύ μεγάλο. Ε, ε, η τεχνολογία του είναι, στηρίζεται σε έρευνα εχμής και είναι πηγή θέσεων εργασίας και εργασίας για την γενικότερη, την ευρύτερη ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό γίνεται τώρα, δεν θα γίνει το 2050 ή 70. Επίσης είναι μακράς πνοής απάντηση στη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιματική αλλαγή και δεν μπορούμε να περιορίσουμε το έργο μας εξετάζοντας μόνο τα σημερινά θέματα. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, διευκρίνησε πολλά σχετικά με τον Ίτερ όταν πέρσι δημοσιεύσαμε μια ανακοίνωση που την ανέφερε και ο κύριος Ζανονάτο στην ε, παρεμβασή του, όπου κάνουμε σαφέστατη ανάλυση της τωρινής κατάστασης και του τι χρειάζεται για το μέλλον. Δηλαδή ε, χρηματοδοτικούς πόρους για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές και πέραν αυτού. Μέχρι ε, αρχίσουν να λειτουργούν όλα 100%. Η πρόταση της Κομισιόν είναι 6, δις και 70 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις που ε, ετέθησαν από την κυρία Ριβάζη από τους Πρασίνους. Πρώτον, πότε θα συνδεθεί στο δίκτυο ο ΙΤΕΡ. Δεν είναι σχεδιασμένος για να συνδεθεί στο δίκτυο. Ο ΙΤΕΡ θα αποδείξει την επιστημονική δυνατότητα της σύνδεξης ως ενεργειακού μέσου. Αυτό σημαίνει ότι θα παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι εισραίει σε αυτόν για αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό θα κάνει ο ΙΤΕΡ. Θα υπάρξουν αρκετά βήματα που θα χρειαστεί να στηρίζονται στην εμπειρία του ΙΤΕΡ και που θα ε, αποδεικνύουν ε, την πολιτική μας. Και υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την κατασκευή του μηχανήματος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τον παροπλισμό του. Ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ταμείο, είναι ξεκάθαρο αυτό, που θα χρησιμοποιηθεί για τον παροπλισμό του μηχανήματος. Και σας θυμίζω πράγματι ότι όντως το μηχάνημα ε, δημιουργεί ενεργά υλικά, αλλά αυτά είναι τελείως διαφορετικά υλικά από ότι αυτά που δημιουργούνται στους συμβατικούς αντιδραστήρες σύνδεξης και έτσι οι τεχνικές για το χειρισμό αυτών των υλικών είναι συγκριτικά απλούστεροι όπως και η διάρκεια ζωής των ε, υλικών που προκύπτουν Σταματώ εδώ και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Και ο κύριος Μαρινέσκου, ο εισηγητής μας, θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια απάντηση στην ερώτηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χώρα υποδοχής. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ χώρας υποδοχής και ΙΤΕΡ και τη σύνδεξη για την ενέργεια, του F4 Energy. Η Γαλλία είναι η χώρα υποδοχής, αλλά θέλω να το επισημοποιήσω γιατί όλα αυτά στηρίζονται σε άτυπες συμφωνίες. Γι' αυτό το έβαλα. Αυτό ετούμε στην έκθεση. Αυτά μόνο και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Οι συνάδελφοι του Ήτρε θέλουν να επισκεφτούν τον χώρο και το project αυτό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη και όλοι μας θα έλεγα συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να είμαστε καινοτόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η καινοτομία πάντοτε συνεπάγεται ρίσκο. Χωρίς ρίσκο δεν γίνεται καινοτομία το να σταματήσουμε όλο αυτό το ε, εγχείρημα ε, θα σημαίνει ότι ε, καταργούμε κάθε καινοτομία στην Ένωση. Οπότε δεν υπάρχει εναλλακτική για να το πούμε απλά. Μόνο μπροστά μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι διεθνές το πρόγραμμα αυτό και πρέπει να είμαστε σε ηγετική θέση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11 Οκτωβρίου, ψήφο στην Ήτρα 21 Νοεμβρίου, Πάμε στο επόμενο σημείο, το 12. Ε, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής έχουμε σχέδιο ε, έκθεσης. Ο συνάδελφος Ζωάο Φερέιρα από την ΚΟΕ είναι ο εισηγητής μας και πρόκειται για την προετοιμασία του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 29 Μαΐου ο νέος ενιαίος κανονισμός για τα δύο Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής ε, εντοπίζουν συγκεκριμένους στόχους και στήριξη και για τα δύο ταμεία, συμπεριλαμβάνοντας ε, και δραστηριότητες μη επιλέξιμες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει η δυνατότητα τα, να εντάξουμε σημαντικά θέματα ε, για την Ήτρε είτε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είτε το Ταμείο Συνοχής γενικότερα. Λοιπόν, ο συνάδελφος Μιγγέλ Βιέγκα αντικαθιστά τον κύριο Ζωάο Φερέιρα από την Γκουε να αρχίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Εξηγώ γιατί βρίσκομαι εδώ. Γιατί ο συνάδελφος κύριος Φερέιρα δεν μπορούσε να έρθει λόγω άλλων υποχρεώσεων στην Πορτογαλία. Έπρεπε λοιπόν να έρθω εγώ και θα διαβάσω τις σημειώσεις του μόνο. Ε, μετά το έργο που ανέλαβε ως εισηγητής. Η βασική προϋπόθεση που χρησιμοποιεί ο κύριος Φερέιρα είναι η διατήρηση της βασικής λειτουργίας της πολιτικής συνοχής, η οποία πρέπει να είναι η μείωση ε, δαφικών και κοινωνικών ασυμμετριών και θα καταπολεμεί τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή πρέπει να είναι η έμπνευσή μας στην πολιτική συνοχής και πιο συγκεκριμένα ε, τον προσανατολισμό των δύο ταμείων επίσης. Ε, έχουμε καταλήξει ότι οι διαβουλευόμενοι θεωρούν ότι η μείωση των διαπεριφερειακών ανισορροπιών είναι πολύ σημαντική και μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Οπότε αυτό είναι το αφετηριακό σημείο και αναπόφευκτα. Έτσι πάμε σε ένα αρνητικό συμπέρασμα. Μιλάμε για κανονισμό εδώ, ο οποίος θα ε, προβλέψει σημαντική 10% μείωση στα ταμεία και 45% στο Ταμείο Συνοχής. Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα νέα, τα οποία υπονομεύουν τους βασικούς μας στόχους. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί στην πράξη να μιλάμε εδώ για διπλή μείωση, Πρώτον, μία ποσοτική μείωση, γιατί τα, ε, όλα τα ποσά περικόπτονται, αλλά και ε, ε, να έχουμε και ένα κλάδεμα στους στόχους και μείωση της δυνατότητας επιλογής ε, από τα κράτη-μέλη, την ευρύτητα των επιλογών που είχαν. Αυτές είναι οι ιδέες που προωθούμε και εκφράζουμε και στις τροπολογίες. Εγώ επικεντρώνομαι στην συνοχή για να μειώνονται οι εδαφικές ανισότητες και παράλληλα η προσπάθεια είναι να υπάρχει αρκετή ευελιξία ε, για να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά της θεματικής συγκέντρωσης. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα να γίνονται διαπραγματεύσεις αναχώρα για να βγούμε από αυτό το ζρουλομανδία, αν θέλετε που μπορεί να είναι η θεματική συγκέντρωση ώστε τα κράτη-μέλη να διοχετεύουν τα ε, κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κατά τη γνώμη τους. Και βέβαια οι προϋποθέσεις και οι ανάγκες διαφέρουν από, μεταξύ περιφερειών. Εγώ θα αναφέρω κάποια βασικά σημεία που καλύπτουν οι τροπολογίες μας και αφορούν ε, καθολικές ε, δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ε, βιώσιμη κινητικότητα υψηλής ποιότητας στις περιφέρειες και διαπεριφερειακά και ε, χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Στους σιδηροδρό... Ε, πρόθεση σιδηροδρόμων, παραδοσιακούς τρόπους συμμετοχής στην αξιακή αλυσίδα, η επαναβιομηχανοποίηση περιοχών που επλήγησαν από βιομηχανική παρακμή είναι πολύ σημαντική γιατί χωρίς θέσεις εργασίας δεν υπάρχει συνοχή και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οικονομικές ασυμμετρίες χωρίς να προωθήσουμε την απασχόληση σε αυτές τις ε, περιφέρειες ανάπτυξη ικανοτήτων και υποδομών για την καλύτερη δυνατή χρήση της γαλάζιας οικονομίας, ε, στέγη, ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών με ταυτόχρονο σεβασμό του περιβάλλοντος, ε, η πολιτική στέγη... Ε, είναι πολύ σημαντική και τέλος αλλά πολύ σημαντικό οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Γιατί πιστεύομαι ότι η αντιμετώπιση του σήμερα είναι απαράδεκτη. Αυτή είναι και η πρώτη μας πρόταση. Ο Ζωάο Φερέιρα θέλει να ευχαριστήσει τη Γραμματεία για την υποστήριξή της και ο Ζωάο προφανώς θα είναι στη διάθεσή σας και ε, έτοιμος να συνεργαστεί με τους κοιόδους για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, είναι σημαντικές και οι τροπολογίες για να υπάρξει χρηματοδότηση. Θα μιλήσουμε τώρα, θα, δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ράτκε εκ μέρου του ΕΛΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, τη απουσία του κυρίου Φερέρα θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. για την θέση που εξέφρασε. Εγώ θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για αυτό το θέμα, που είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εκφράσω επίσης την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ. Γιατί προέρχομαι από ε, το Ρούρ που είναι που ιστορικά ε, χαρακτηρίστηκε από την ε, Χαλιβουργία. Είδαμε πόσο πολύ μειώθηκε η απασχόληση στον τομέα αυτό, όχι μόνο στη δική μου περιφέρεια, αλλά και σε άλλες γερμανικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μια διαρθρωτική αλλαγή ε, αρκετά σημαντική. Πρέπει να υπάρξει και συνεργασία αλλά και συντονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλές φορές έχουμε δει παραδείγματα ομαλής αλλαγής, αλλά έχουμε δει περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες η απασχόληση χάνεται στον βιομηχανικό τομέα και αντικαθίσταται από ε, απασχόληση στον ψηφιακό τομέα ή στον τομέα της πληροφορικής ε, με πολύ χαμηλούς μισθούς, κάτι λοιπόν που σημαίνει ότι η οικονομική βάση υφίσταται μία διάβρωση, για να το πω έτσι. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες διαρθρωτικά περιοχές θα μπορέσουν να εξακολουθούν να επωφελούνται από τις ενισχύσεις αυτές. Έχουμε μια δραστηριότητα ε, του τύπου πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στους πέντε πολιτικούς στόχους που αναφέρονται στο γενικό κανονισμό θέλω να τονίσω με θετικό τρόπο ότι δεν αναφέρεται μόνο σε επίκαιρα σημερινά θέματα δηλαδή, αλλά μπορούν να το δουν ε, όλοι ότι προσπαθούμε να έχουμε και υλοποίηση του πυλώνα για τις κοινωνικές ανάγκες και είχε πει και ο κύριος Γιούγκερ άλλωστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι σωστό και συνεπές σε αυτό το σημείο να αναφέρεται. Και τέλος και το θέμα της ε, ε, ενσωμάτωσης των μεταναστών, ένα θέμα που δίχαζε μέχρι τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκείνοι που λένε ότι θα βοηθήσουμε στο προσφυγικό, με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί ε, τρόπος ε, για την ένταξη των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε για όλες τις παρατηρήσεις. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ρούπερτ Μάθιους, εξ ονόματος της ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την, ε, το σχέδιο έκθεσης. Μπορούμε να στείλουμε γρήγορα οδηγίες στη Ρέτζη για τα ψηφιακά θέματα και την ενέργεια. Ε, το θέμα είναι σημαντικό. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντική για όσους έχουν ανάγκη. Είμαστε υπέρ της ε, πρότασης της Κομισιόν ε, η καθαρή ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η καινοτομία είναι τα πιο σημαντικά. Δεν έχουν υπερτονιστεί. Εναρμόνιση κανόνων χρηματοδότησης, μείωση διοικητικών ε, φόρτων, ε, καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι στις προτάσεις. Συμφωνούμε με τις προτεραιότητες, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν διακριτική ευχαίρεια να προσαρμόζουν τις δραστηριότητε. Ε, χρειάζεται απλούστευση ε, περισσότερη. Ε, νομίζω ότι είναι καλή η ευελιξία που εισάγεται, δηλαδή τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερα κονδύλια για τις προτεραιότητες. Επίσης να αντιμετωπίζουν τους στόχους εκπομπών σε σχέση με την πράσινη πράσινες εκπομπές Επίσης, ε, οι περιοχές ε, των οποίων ο πληθυσμός μειώνεται χρειάζονται επίσης κονδύλια και αυτό είναι σημαντικό. Όμως, ε, οι κρατικές ενισχύσεις και κρατικοί κανόνες θα ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Κατανοούμε τους στόχους του εισηγητή, αλλά νομίζω ότι αν έχουμε στόχους <clears throat> στέγης και πλήρους απασχόλησης, δεν θα μπορέσουμε με αυτό να ε, αναζωογονήσουμε την οικονομία. Ελπίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα μπορέσει να επηρεάσει τον τελικό κανονισμό. Προσβλέπω σε μια συνεργασία προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αντακαταστήσετε τον κύριο Ρικέ ε, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριο Ρικέ σήμερα το πρωί γιατί έχει πάρα πολλέ εκθέσει ε, στην Επιτροπή Μεταφορών ε, και συζητιούνται την ίδια στιγμή. Θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την ε, περιεκτική του έκθεση. Συμφωνεί ως προ τον τονισμό ενός από τους βασικούς στόχους των, των ταμείων, δηλαδή τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ ε, των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει την οργάνωση σε θεματικές ενότητες, ε, θεωρεί ότι είναι μία αποτελεσματική διάκριση. Συμφωνεί με τον εισηγητή ότι τα διάφορα ποσοστά ε, των συγκεκριμένων ε, στόχων θα έπρεπε να μειωθούν κατά τη. Επίσης, ε, ο κύριος Ρικέ θεωρεί ότι κάποιες από τις τροπολογίες πηγαίνουν πολύ μακριά. Αντιθέτως, θεωρεί ότι κάποιες δεν είναι αρμοδιότητα της Ήτρε, παρά το ότι αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Ο κύριος Ρικέ και θα υποβάλει τροπολογία όσον αφορά το, το 20%, τη μεταφορά 20% από το ERDF στο ECF, από ένα σύνολο 200 δις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ε, στις υποδομές του ε, συνδέοντας την Ευρώπη, του CEF, ε, να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που φάνηκαν να είναι πολύ αποτελεσματικές. 10 δισεκατομμύρια ευρώ μεταφέρονται τώρα λογικά στο συνδέοντα την Ευρώπη από 41 δισεκατομμύρια συνολικά. Ελπίζεται, ο, ε, εκφράζει την υποστήριξή του στην έκθεση και ελπίζει να ε, συζητήσει με τον εισηγητή ε, σύντομα. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν μέλο τη Επιτροπή Παρακολούθηση για, για τα προγράμματα του στόχου 1 τη δεκαετία του 90, όταν ήμουν τοπική σύμβουλο. Ήταν ευρωπαϊκά χρήματα αυτά που βοήθησαν ε, στη μεταμόρφωση των πιο ε, απομακρυσμένων περιοχών και ακριβώ ε, η σύνδεση του CF με το ERDF ήταν πολύ σημαντική γιατί αφορούσε την εκ νέου κατάρτιση και τα χρήματα είχαν άμεση σχέση και με την παιδική φροντίδα γιατί και επέτρεπαν στις γυναίκες να συμμετέχουν και δεν θα ήθελα να αναφέρω και πάλι αυτά που είχα πει στο Λίβερπουλ ε, τότε αλλά πρέπει να πω ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι αυτά που μεταμόρφωσαν την πόλη του Λίβερπουλ το, το θέμα αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι να ε, γνωστοποιούνται οι αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι περιφέρειες είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Είναι διαφορετικό το κοινωνικό και οικονομικό σημείο αφετηρίας και η τοπική εμπειρογνωμοσύνη που προέρχεται από όλους τους φορείς και κατά το σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο κράτους μέλους. Πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο και με ε, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Τεχνικής ω παρατήρηση για το μέλλον. Καταλαβαίνω ότι θα προτιμούσατε περισσότερη ευελιξία στην ε, απόφασή μας, αν κατάλαβα καλά την παρέμβασή σας. Ο κύριος Κόχιτσεκ επίσης θέλει να πει, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η τσεχική δημοκρατία λόγω της γεωγραφικής της διαμόρφωσης έχει πολλές ε, μεθοριακές περιοχές οι οποίες έχουν καθυστερήσει Επίσης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαρθρωτικά προβλήματα επειδή υπάρχει μεγάλη ανεργία λόγω του ότι δεν γίνεται εξόριξη άνθρακα πλέον. Το επίπεδο της ε, ανάπτυξης των περιφερειών πρέπει να προσεγγίσει το ένα το άλλο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις μεταρρυθμίσεις ε, που, χρειαζο... που συζητούμε σήμερα. Χρειαζόμαστε τη διευκόλυνση συνθέοντας ε, την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε διάφορες μορφές ε, διασυνοριακής συνεργασίας. Πρέπει να αυξήσουμε την ευελιξία όσον αφορά τη χρήση των ταμείων αυτών. Και επίσης πρέπει να απλοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διοικητικές διαδικασίες. Στη Τσεχική Δημοκρατία οι περισσότερες περιφέρειες που χρειάζονται ε, που πρέπει να καλύψουν την καθυστέρησή τους στην οικονομική είναι ε, περιοχές απομονωμένες ε, της υπαίθρου που έχουν πολλά προβλήματα αντιμετώπισης όλων αυτών των δύσκολων διοικητικών διαδικασιών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μόρι Τζίλεντ, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για τη δουλειά του. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 αφορά ε, τη δημιουργία μιας πολιτικής υποστήριξης ε, που είναι συντομότερη, απλούστερη και πιο εύκολη στην εφαρμογή της. Ε, είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς της διατύπωσής μας και του επίπεδου λεπτομέρειας που θελήσαμε να επιτύχουμε όσον αφορά λοιπόν το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα ευέλικτο ε, περιεχόμενο. Έχουμε πέντε στόχους, ε, πέντε κεφάλαια που συγκεντρώνουμε γύρω από 20 στόχους σε σχέση με τις 11 θεματικές ενότητες και ε, σε 40 επενδυτικές προτεραιότητες Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη ευελιξία για τα προγράμματα των περιφερειών. πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ε, την, ε, τη θεματική αυτή συγκέντρωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο στόχος της, η εστίαση της είναι να υπάρξει μία σχέση μεταξύ της συνολικές ε, σφαιρικές πολιτικές και προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωση και ε, του πού πηγαίνουν τα χρήματα των ταμείων συνοχής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο στόχος μας ε, εστιάζεται κυρίως σε μία χαμηλής περιεκτικότητα σε άνθρακα η οικονομία και στις σχετικές δαπάνες. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν, αλλά δεν θέλουμε δαπάνες πολλές σε πολύ διαφορετικές προτεραιότητες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μεωθεί ο συνολικός αντίκτυπος και το αποτέλεσμα της πολιτικής συνοχής στο σύνολό της. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 6 ε, της, επιτροπής, ε, της πρώτας επιτροπής όσον αφορά τον αποκλεισμό από τα ε, κονδύλια αυτά συνδέεται με άλλες πολιτικές, σε άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήταν πολύ αντιπαραγωγικό αν δημιουργούσαμε πολιτικές από τη μία και από την άλλη ξοδεύουμε χρήματα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από το άρθρο 6. Και θα ήθελα Συμπερασματικά να πω ότι άκρος περιφερειακές ε, περιοχές ε, είναι μεγάλης προτεραιότητας περιοχές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει χρηματοδότηση που προβλέπεται υπό την τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, επιπλέον ευελιξία στο, στην πρόταση έχει προβλεφθεί για να ληφθεί υπόψη τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις προτάσεις σας και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα σύγκλησης πάνω σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν βρει την σωστή τους έκφραση στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Και βεβαίως εμείς μπορούμε να ε, ε, να προχωρήσουμε ε, όσον αφορά τα ε, σημεία αυτά ε, και να βρούμε κοινή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, 10 Οκτωβρίου για τις τροπολογίες, 21 Νοεμβρίου στην Ήτρε και στην Περιφερειακή, στη Ρέγγι, στις 3 Δεκεμβρίου οι ψηφοφορίες. Σημείο 13 της ημερησίας διατάξεως. Θέσπιση προγράμματο έρευνα και κατάρτιση τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια για την περιοδο 2021 2021-2025 με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία ορίζων Ευρώπη. Η συνάδελφος Μια Πέτρα Κούμπουλα Νάτρη θα έχει το λόγο. Όπως σας είπα, αυτό αποτελεί τμήμα του προγράμματος πλαισίου για τη, το, τη γενοτομία ορίζων ε, Ευρώπη ε, και ε, αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος με κάποιες προσαρμογές. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζητήθηκε διαβούλευση όσον αφορά αυτήν την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 7 της Συνθήκης Ευρατόμ. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την εισηγήτριά μας, κυρία Μια Πέτρα Κουμπούλα Νάτρη, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό είναι τμήμα του προγράμματος έρευνας Horizon Europe για το οποίο είχαμε μια πολύ καρποφόρα συζήτηση ε, χθες. Ε, ε, είναι ένα πρόγραμμα με μεγάλη χρηματοδότηση. Σήμερα μιλήσαμε για θέματα τα οποία σχετίζονται με τα πυρηνικά και για το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο εντάσσεται στις ε, ε, προσπάθειες που κάνει η καταβάλη Ευρώπη στον τομέα αυτό. Έχουν γίνει ε, μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τα παλαιότερα προγράμματα και θα πρέπει να συνεχιστούν στο επόμενο πρόγραμμα. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι πρέπει ε, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο από πιο κοντά αυτή την αυτό τον τεχνητό διαχωρισμό Ευρατόμ και Horizon Europe έτσι ώστε ε, το ε, ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρατόμ να συμπεριληφθεί απολύτως και στις διαδικασίες βάσει των οποίων προβλέπεται διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα έρευνας κατάρτισης τη το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon ε, Ευρώπη. Ε, ξέρω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες νομοθετικές τροποποιήσεις, αλλά μπορούμε να τις προετοιμάσουμε. Σε γενικές γραμμές η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά την Ευρατόμ ε, είναι καλοδεχούμενη. Γενικώ ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει το πρόγραμμα να αναπτυχθεί μας βρίσκει σύμφωνο, πούμε ε, ε, να είναι επιλέξιμοι για τις ε, δράσεις του προγράμματος Μαρή Κυρί, Μαρής Λαντόφσκη, και οι ερευνητές του προηγούμενου προγράμματος. Επίσης, άλλωστε το πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon Europe έχει λάβει πολλά στοιχεία από τις προτάσεις της Κομισιόν. Επίσης, γνωρίζουμε ότι είναι τρία τα κύρια στοιχεία του προγράμματος, θέματα τα οποία αφορούν την πυρηνική ενέργεια, την ασφάλεια και την προστασία των πυρηνικών ε, το κοινό κέντρο ERC, καθώς επίσης ε, και το θέμα της ε, σύνδεξης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μεγιστοποιήσουμε την επίπτωση της έρευνας, ενώ θα, ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ε, ε, υποχρεώσεις ε, για την κλιματική αλλαγή έτσι όπως έχουν αναλυφθεί στο Παρίσι θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, δούμε και το ενεργειακό μείγμα των ε, χωρών και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να προχωρήσουμε στην απανθρακοποίηση του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δηλαδή την μείωση, την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ανθρακούγες εκπομπές στο σύνολό του και βεβαίως ζωτική σημασία είναι η ασφαλή λειτουργία των υφισταμένων μοντέλων αντιδραστήρων καθώς επίσης και η προετοιμασία των νέων τεχνολογιών. Ε, ε, ο πυλώνας της έρευνας όσον αφορά την ασφάλεια ε, της σύνδεξης είναι ένα σημαντικό στοιχείο του ERC και εδώ εμείς προτείνουμε και κάποιες επιπλέον, κάποια επιπλέον κονδύλια. Το ERC αποτελεί εξαιρετική βάση. Το ζήτημα είναι χρειαζόμαστε περισσότερες, περισσότερη χρηματοδότηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ε, μεγαλύτερη ασφάλεια ε, στον πυλών αυτό. όσον αφορά την ε, συνεχίση της χρηματοδότησης για την έρευνα, για τη σύνδεξη, βεβαίως είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να συνεχίσει. Από την άλλη πλευρά η χρηματοδότηση ήταν θα έπρεπε να ήταν ίσως διαφορετική τώρα το κατά πόσον θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί ε, η σύνδεξη και στο παρελθόν ή ήδη από το παρελθόν δεν ξέρω εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνει εγώ δεν προτείνω καμία αλλαγή όσον αφορά αυτόν τον πυλώνα βεβαίως χρειάζονται επενδύσεις για την ανάπτυξη ε, της ε, έρευνας για την σύνδεξη και ε, είναι γεγονός ε, ότι για το υφιστάμενο πρόγραμμα η Ολομέλεια είχε με μεγάλη πλειοψηφία ε, αποδεχθεί την συνέχιση της χρηματοδότησης και αυτό θα πρέπει να το δούμε και για το μέλλον όσον αφορά τη σύνδεξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος για τις παρατηρήσεις σας. Σκιώδης εισηγητές. Η κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ από πλευράς ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. Έχουμε εδώ ένα πρόγραμμα το οποίο είναι θεμελιώδους ε, σημασίας ε, για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα για την πολιτική μου ομάδα. Η η ενέργεια από, που προέρχεται από πυρηνική ενέργεια μας έχει απασχολήσει. Έχουμε βέβαια ταυτόχρονα και στόχο της μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών ε, στην ε, Ευρώπη. Ε, θέλουμε απαλλαγή μακροπρόθεσμα του ενεργειακού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές στο σύνολό του ε, ε, και εδώ έχουμε επομένως πολλές δυνατότητες που μας παρέχονται από μια ε, πολύ από μια πολύ καινοτόμα διαδικασία. Άλλωστε και το θέμα της σύνδεξης που μας απασχόλησε στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας από σύνδεξη του προγράμματο ITER έχει δείξει το δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να έχουμε και χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα αυτό ε, διότι ο αντίκτυπος μπορεί να είναι πολύ σημαντικό σε πολλούς τομείς στην υγεία με την ραδιοπροστασία ε, των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν όλες οι δυνατές Συνέργεια στον τομέα αυτό. Επίσης ε, έχουμε ένα τεράστιο διακύβευμα όσον αφορά την ασφάλεια, ασφάλεια συστημάτων, ασφάλεια ε, ε, των ατόμων. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία του προγράμματος είναι πολύ σημαντικά. Εξού και η ανάγκη για πολύ σημαντική χρηματοδότηση αλλά και δυνατότητα ευελιξία ανάμεσα στις διάφορε στρατηγικέ προτεραιότητε. Υποστηρίζω την εισηγήτρια στην πρότασή της όσον αφορά τη ραδιοπροστασία και την ε, ε, σύνδεξη που θα πρέπει ε, να τύχουν μεγάλη χρηματοδότηση, χωρίς όμως να λησμονήσουμε και την έρευνα ε, ε, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν, ε, για τις χάσεις, συγγνώμη, δεν θα πρέπει βεβαίως να ξεχάσουμε και την σύνδεξη που είναι πάρα πολύ σημαντική, επομένως σημαντική χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου προγράμματος, γιατί είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κοχέτσικ από Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την συνάδελφο, καθώς επίσης, την συνάδελφο εισηγήτρια, καθώς επίσης και την ε, κυρία Γκροστέτ για την υποστήριξη του προγράμματος. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν αναφέραμε όμως ε, αναφέρομαι στην προώθηση και την υποστήριξη κατάρτισης ακόμα και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή δημιουργούμε μία ολόκληρη γενιά που βγαίνουν από αυτά τα σχολεία και από αυτά τα πανεπιστήμια που ακούν διαρκώς ε, ε, ε, πράγματα κατά της πυρηνικής ενέργειας. Λείπει λοιπόν το κατάλληλο προσωπικό, αλλά δεν είναι δυνατόν στον τομέα αυτό να χρησιμοποιηθεί προσωπικό που δεν θα έχει λάβει την απαραίτητη κατάρτιση δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς ε, το πυρηνικό υλικό εάν δεν είναι υψηλότερα καταρτισμένος. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Επίσης ε, θα πρέπει ε, να αναφερθούμε οπωσδήποτε στον, στην χρήση πυρηνικών από την πυρηνική τεχνογνωσία, σε πάση περιπτώσει, στην ιατρική ραδιοτεχνολογικό, ιατρικό υλικό για την αντιμετώπιση ασθενειών και αυτό πρέπει να το πούμε με έντονο τρόπο. Τρίτον, ε, ε, είναι και ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και στα πλαίσια της έκθεσης ε, του συναδέλφου Κουλούμπου Σεφ. Πρόκειται για την έρευνα, για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα ε, υψηλά ή ασθενώς ραδιοενεργά ε, υλικά στα πλαίσια του παροπλισμού <clears throat> ε, των εγκαταστάσεων. Ε, είτε μιλάμε για κοβάλτιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ε, ιατρική, είτε μιλάμε για άλλα υλικά. Ε, πραγματικά θα πρέπει να τα αναφέρουμε στο μέλλον, γιατί πρόκειται για στοιχεία στα οποία και τομέα των οποίων μπορούμε να είμαστε ηγέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ταμπουράνο, ε, εξ ονόματος ε, του FDD. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, συμμεριζόμαστε το αίτημα της εισηγητρίας για μεγαλύτερη ανάμεξη του Κοινοβουλίου και επίσης ε, το αίτημα να συνδυαστεί ε, το ορίζον Ευρώπη με τις ε, <clears throat> πολιτικές προτεραιότητες. Όμως, εμείς θεωρούμε ότι η έρευνα στον τομέα της, της πυρηνικής ενέργειας στη, δεν θα πρέπει να οδηγήσει με, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να οδηγήσει στην παράταση ζωής παλαιών ε, εγκαταστάσεων. Έχουμε αυτή τη στιγμή 138 αντιδραστήρες ε, στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια δαμόκλειο σπάθη η οποία επικρέμεται ε, των κεφαλών των Ευρωπαίων πολιτών στο, σε αυτό το κοινό μας σπίτι ε, ε, όπου πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε χρήματα έτσι ώστε να παροπλιστούν αυτοί οι, οι σταθμοί. Δεν είναι δυνατόν, λέω, να μην χρησιμοποιούμε χρήματα για την πραγματική ασφάλεια και για το πραγματικό τελειωτικό κλείσιμο, οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της και ε, στην αντιμετώπιση των ραδιονεργών αποβλήτων ε, που ε, ακόμα υπάρχουν και διακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουν τεράστιο κύκλο ζωής. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεσοβαλιέρα, εξ ονόματος του ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εμείς ε, υποστηρίζουμε τους διαφορετικούς στόχους της Ευρατόμως επίσης και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική μείωση του προπολογισμού που μας λείβει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα ενεφοδιασμού σε ενέργεια, προβλήματα για την υγεία, όπως επίσης και για το περιβάλλον με 1,67 δισεκατομμύρια που προβλέπονται για πέντε χρόνια. Το πρόγραμμα προβλέπει 334 εκατομμύρια κατ' ενώ ήταν 418 για το 2002 ε, ε, με 2007 και ακόμη, περισσότερο ήταν την, ακόμη λιγότερο ήταν την επόμενη περίοδο. Ε, δεν επιτρέπει λοιπόν να υπάρξει αξιοποίηση του δυναμικού της χάσης. ακόμη και αν δεν υπάρχει ελληνική εγκατάσταση σε μία χώρα είναι πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη. Ε, είμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση της ε, ε, συνθήκης της Ευρατών. Παρόλα αυτό θα ήθελα να πω ότι η πυρηνική ενέργεια, ναι, μεν είναι μια ενέργεια που μπορεί να μειώσει τη χρήση του άρθρακα, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει την έρευνα για τη σχάση που είναι σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματο. Συμφωνούμε ε, με τους στόχους για τη σχάση, όμως έχουμε μια μικρή αντίρρηση όσον αφορά ε, την, ε, το γεγονός ότι πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο κάθε φορά στην αναθεώρηση του προγράμματος, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις για ένα ε, θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνας θα πάρει το λόγο, ο κύριος Σάιλτ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ε, τους αξιότιμους ευρωβουλευτές ε, που συμμετείχαν σε αυτήν την μάλλον ε, θετική συζήτηση της, πρό... της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν και η πρώτη συζήτηση. Υπάρχει μια συνένεση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση μετά από την καταστροφή του ε, της Φουκισάμα ε, για την αναθεώρηση της Ευρατόμ ε, με σκοπό την προστασία από την ακτινοβολία και την ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο το είπατε. Το όλα αυτά στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματός μας για τη σχάση. Εμείς επικροτούμε την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις που κάναμε για το πρόγραμμα Ευρατόμ ε, ειδικότερα ε, μα ενθαρρύνει η ισχυρή πλειοψηφία ε, υπέρ του, της αναθεώρησης του προγράμματος μετά το 2019-2020. Υπάρχουν κάποιες διοργανικές, υπάρχουν κάποιες κάποιοι διοργανικοί, περιορισμοί, αλλά χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως που αναλάβατε την πρωτοβουλία να γνωμοδοτήσετε για ένα τέτοιο κείμενο και Θέλουμε να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε μαζί σας τα διάφορα ζητήματα. Η πρότασή μας ε, ε, συνεχίζει ουσιαστικά, προσπαθεί να συνεχίσει την πρόσφατη επιτυχία της ε, κατάρτισης υπό την Ευρατόμ. Θα ήθελα να τονίσω μερικά στοιχεία υπό το φως της συζήτησης που μόλις άκουσα. Καταρχάς ότι σκοπό έχουμε όντως να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και απλουστευμένη παρουσίαση των συνολικών στόχων για να εξασφαλίσουμε μια καλή σύνδεση μεταξύ του, των εμέσως χρηματοδοτούμενων ερευνητικών δραστηριοτήτων και της εξαιρετικής δουλειάς των συναδέλφων του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Θα έλεγα η πρόταση τροπολογίας, τροπολογιών βέβαια στην ε, έκθεση της εισηγήτριας που θα ήθελε αναθεώρηση του προπολογισμού θα μας δημιουργούσε μερικά προβλήματα πρέπει να πω γιατί η πρότασή μας προσπαθεί να εξεύρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, συνιστοσών και ε, Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει έτσι ένας εναρμονισμένος συντονισμός. Αυτό θα θέλαμε να το συζητήσουμε περισσότερο. Από την άλλη, άλλα σημεία που κατέδειξε η συζήτηση αυτή πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της επόμενης γενεάς ε, ερευνητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το σημαντικό επίπεδο δραστηριότητας και διανοητικής ηγεσία στον τομέα αυτό, ειδικότερα με τη συμπερίληψη των ε, πυρηνικών ε, ερευνητών ε, στις δράσεις Marie Curie. Η συγκήτρια σωστά είπε ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητη η συνοχή μεταξύ του ορίζοντα, 2000, του ορίζοντα Ευρώπη και της Ευρατόμ ο συνάδελφος Βαντελμπέργκε που εχθές ε, ήταν εδώ σας είπε ε, ότι για πρώτη φορά έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις μας ε, για το νομικό κείμενο μια σαφή νομική βάση για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο προγραμμάτων που πιστεύουμε ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, σεβόμενη βεβαίως τη βάση, την τη διαφορά ε, μεταξύ ε, της ε, συνθήκης Ευρατόμ και του ορίζοντα Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την ιονίζουσα ακτινοβολία, Μέχρι τώρα ό,τι έχουμε κάνει αφορά τον ιατρικό τομέα θα θέλαμε να το επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς όπως, άλλους τομείς, όπως τη βιομηχανία, το περιβάλλον και την ασφάλεια. Εν ολίγης, αυτή η πρώτη συζήτηση για μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για να καταλάβω τα ζητήματα που απασχολούν τους αξιότιμους ευρωβουλευτές και θα τα λάβω υπόψη μου, θα τα ξανασυζητήσουμε κατά τη συζήτηση των ε, τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Κουμπούλα Νάτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ χαρά θα συζητήσω και τις τροπολογίες μαζί σας αφού θα τις έχω επεξεργαστεί με τους κοιόδης συζητητές. Ε, είναι σαφέστεροι οι στόχοι και έχουν συμπεριλάβει την ανάπτυξη της τεχνολογίας για τον παροπλισμό. Ε, το επικροτώ αυτό, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο παροπλισμός πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον τομέα. Δεν είναι δυνατόν πάντοτε με δημόσιο χρήμα να χρηματοδοτείται, αυτό το λέω. Ε, γιατί προφανώς ο παροπλισμός χρειάζεται γνώση όσον αφορά στην ασφάλεια. Και θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό τμήμα του προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μία Πέτρα. Τροπολογία, τροπολογίες μέχρι την 5η αυτής της εβδομάδας, 11 Οκτωβρίου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ξανασυναντηθούμε στις 2.30. και Και αυτή είναι η προθεσμία μας ε, για το μεσημεριανό γεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λίγες ώρες.